να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Τέλεια, γιατί ε, τώρα στην ε, ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση Αντρέα Γκιούρκ για τη συνέχεια που δόθηκε στα εθνικά σχέδια δράση για την ενεργειακή απόδοση. Μια πρώτη αξιολόγηση. Το λόγο έχει ο εισηγητή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Επίτροπε. Η ε, κρίση του Ιανουαρίου είχε μια θετική επίπτωση διότι σε όλα τα κράτη-μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλήσαμε ε, για ενεργειακή απόδοση, για εναλλακτικά σχέδια, για το μελλοντικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας. Αλλά η ενεργειακή αποτελεσματικότητα είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε προσέξει επαρχώς και γι' αυτό χαίρομαι ότι κατόπιν της ε, ε, εκθέσεως μπορούσαμε να συζητήσουμε ε, το θέμα αυτό την περασμένη εβδομάδα ε, διότι με την ενέργεια μπορεί κανείς να έχει πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Ο κύριος Πίμπαλξ μας είπε ότι χρειάζεται μία νέα ρυθμισή για να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε εύκολα ε, όση, οικονομία, όση ενέργεια χρειάζεται η Ουγγαρία παραδείγματος χάρη για ένα χρόνο. Θα έπρεπε να μειώσουμε την εξάρτηση της Ευρώπης από τρίτες χώρες όσον αφορά τις παραδόσεις ενεργειακών πόρων. Επίσης θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε διότι οι πιο φτωχοί δεν θα πλήρωναν πολύ υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού. Τα μέτρα ε, που έχουν ληφθεί σε επίπεδο ευρωπαϊκών κρατών διαφέρουν. Γι' αυτό και κατόπιν της απόφασης του 2006 κάθε κράτος έπρεπε να παρουσιάσει μία έκθεση σχετικά με την ε, τα προγράμματα του αποδοτικότητας και εξοικονομήσεως ενεργείας αλλά δεν είχαμε καλά αποτελέσματα θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η πορεία που πρέπει να διαγράψουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και εδώ θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σημεία της έκθεσης. Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι πιο επιθετική όταν υπάρχουν καθυστερήσεις υποβολής των στοιχείων. Δεύτερον, πρέπει να δούμε αν τα προγράμματα όντως συνάδουν με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη, διότι συνήθως υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στην, στα χαρτιά και στην υλοποίηση. Επίσης σήμερα η δεν είναι πολλοί οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι μπορούν να επενδύσουν εις ε, την ε, ενεργειακή εξοικονόμηση και τα προγράμματα θα έπρεπε να ε, επεκταθούν. Επίσης θα πρέπει η ενεργειακή εξοικονόμηση να αποτελέσει προτεραιότητα. Πέραν αυτού θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες και είμαι βέβαιος ότι έχουμε το σωστό προσανατολισμό ε, αν υπήρχε πιο αυστηρές προδιαγραφές για την κατασκευή κτηρίων θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα. Επίσης θα χρειαστεί και μία εξρατεία πληροφόρησης γιατί οι καταναλωτές δεν ξέρουν τι σημαίνει ε, ενεργειακή αποτελεσματικότητα δεν ξέρουν τι προσόντα μπορούν ε, να αποκομίσουν από αυτή την προσπάθεια και τέλος μια σκέψη κύριε Πρόεδρε σε μια περίοδο οικονομικής κρίσεως δεν πρέπει να παραμελήσουμε την ενεργειακή αποτελεσματικότητα διότι θα μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να ε, δημιουργήσουμε πολλές θέσεις εργασίας που είναι αναγκαίες όταν υπάρχουν συνεχείς απολύσεις ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος. Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, καλωσορίζω την ευκαιρία να μιλήσω στην Ολομέλεια για την ε, αξιολόγηση της Επιτροπής ε, για τα σχέδια δράσης ε, για την ενεργειακή απόδοση που παρουσιάστηκε στο δεύτερο στρατηγικό πρόγραμμα του Νοεμβρίου και σε προηγούμενες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιανουαρίου του 2008. Ε, μία σύνοψη της τεχνικής αξιολόγησης της Κομισιόν ε, θα παρουσιαστεί σε ένα έγγραφο της Κομισιόν την Άνοιξη. Με αυτήν την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γκύρκ, για τη δουλειά που έκανε και να ευχαριστήσω και την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας Έρευνας και Έρευνας για τις σημαντικές συζητήσεις και τα σχόλια που έκαναν. Τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν ε, τόνισε ξεκάθαρα ότι η ενεργειακή απόδοση είναι η πρώτη προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενεργειακή της πολιτική και είναι ακρογωνιαίο σλήθος της πολιτικής 2020. Τα εθνικά σχέδια δράσης για την ενεργειακή απόδοση παίζουν σημαντικό ρόλο για την πολιτική αυτή. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των ενεργειακών ε, ε, υπηρεσιών βαραίνει με κάποιες υποχρεώσεις τα κράτη-μέλη τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν πώς θα υλοποιήσουν την ευγειακή απόδοση στην πράξη. Η αρχική ε, προθεσμία για τα κράτη-μέλη έλεγε ότι ήταν μάλλον 30 Ιουνίου του 2007. Ξέρετε ότι πολλά κράτη-μέλη όμως καθυστέρησαν δυστυχώς. Ε, ορισμένοι ε, ε, ήταν έτοιμοι τον Ιούνιο του 2008. Έτσι προχώρησε η Κομισιόν σε επιμέρους αξιολογήσεις και έστειλε ε, επιστολές με τα αποτελέσματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Το follow-up ήταν κάποιε διμερεί συναντήσει και κάποια κράτη-μέλη δήλωσαν ότι θα ήθελαν από μόνα του να βελτιώσουν την ε, ενεργειακή τους απόδοση του επόμενους μήνες. Όπως σημειώθηκε από τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε, το πρώτο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση ε, ήταν πολύ σημαντικό Πολλά κράτη-μέλη για πρώτη φορά έχουν ετοιμάσει ευραία σχέδια για ενεργειακές εξοικονομήσεις. Ορισμένοι είπαν ότι κάνουν διατομεακή προσπάθεια, κάτι που είναι απαραίτητο για να εξοικονομήσουν ενέργεια. Με βάση την οδηγία για τις ενεργειακές υπηρεσίες, ε, η ενεργειακή απόδοση θα παίξει περιορισμένο ρόλο. Όμως η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της τον Νοέμβριο και σε πρόσφατες δηλώσεις ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να παίξουν όσο να τον πιο ευρύτερο ρόλο μπορούν. Εμείς θα ετοιμάσουμε ένα νέο σχέδιο δράσης για την εξοικονόμηση ενέργειας που θα ενδυναμώσει τις δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για να εξοικονομήσουν ενέργεια με αποτελεσματικό τρόπο. Στην έκθεσή σας έχετε κάνει κάποιες αναφορές, ε, τονίζετε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να προτείνει ε, δεσμευτικούς στόχους ε, ο στόχος του 20% για τις πρωτογενείς εξοικονομήσεις ενέργειας 2020 είναι μη δεσμευτικό σήμερα, όπως ξέρετε. Όμως πιστεύουμε, εμείς στην Επιτροπή, ότι με το ενεργειακό και κλιματικό πακέτο, καθώς και με τις προτάσεις στο δεύτερο στρατηγικό ε, πρόγραμμα αναθεώρησης, μπορούμε να ε, επιτύχουμε το 20%. Η έκθεση του Γκιουρκ ε, πολύ σωστά λέει ότι η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης είναι πολύ σημαντική. Τα οικονομικά θέματα σε σχέση με την εξοικονόμηση της ενέργειας έχουν αναγνωριστεί από την ε, Κομισιόν στην, ε, στο Ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψη τη 26η Νοεμβρίου και σε άλλε συντονισμένε προσπάθειε που σκοπό έχουν να βοηθήσουν την δημιουργία θέσεων απασχόληση στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, μια και οι επενδύσει στην ενεργειακή απόδοση, ε, ειδικά στα κτίρια, ε, συνδέονται πάρα πολύ με μικρά ε, και καινοτόμα προγράμματα. Για να καταλήξω, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια τη θητείας αυτής της ε, Επιτροπής προσπαθούμε ε, να προωθήσουμε πραγματικά την ενεργειακή απόδοση. Να τονίσουμε τις επενδύσεις ε, σε τεχνολογίες, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και ασφάλεια του ανεφοδιασμού. Η ενεργειακή απόδοση έχει μεγάλη επίπτωση πέρα από τις ενεργειακές πολιτικές. Έχει θετικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία με την ενεργειακή απόδοση θα έχουμε νέε θέσει απασχόληση, θα τονώσουμε την ε, οικονομική ανάπτυξη και θα βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα. Ακριβώ αυτό πρέπει να κάνουμε σε αυτέ τι δύσκολε ε, εποχέ. Πολύ σωστά τα είπατε, κύριε Σιγητά. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Επίτροπε, αύριο στις 10.30 θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή. Τέλος. Έχουμε μια σύντομη παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Μεγγέλης Ράμος για την εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό με τα φώτα που έγινε πριν ήταν υπέροχο. Πρέπει να το επαναλάβετε, να γίνεται πιο συχνά εδώ στην Ολομέλεια.